Λοιπόν, με καθυστέρηση μεν, αλλά αρχίζουμε. Όσοι δεν ε, θέλουν να παραμείνουν για την ακρόαση αυτή, παρακαλώ να αποχωρήσουν ησύχω. Έχουμε λοιπόν το σημείο 15 στην ημερήσια διάταξη, που είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας. Thank you. Thank you for coming. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Thank you. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρέσβη της Ιαπωνίας, τον κύριο Καζού Ακοντάμα, ο οποίος ε, είναι σήμερα μαζί μας για αυτήν ε, την ε, ακρόαση. Οργανώνουμε τη δημόσια αυτή ακρόαση. EU-Japan relations which relates to the Parliament's consent to the EU ε, σχετικά με θέμα την στρατηγική εταιρική σχέση και τη Συμφωνία εταιρική σχέση και Συνεργασίας με την ε, Ιαπωνία. Ε, δεν θα έχουμε την δυνατότητα ε, να ε, έχουμε ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση η οποία σχετίζεται με το θέμα αυτό και επομένως μέσω της ακροάσεως αυτής θα έχουμε την δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω και τους προσκεκλημένους μας ομιλητές, τον κύριο Γκούναρ Βίγκανγκ, ο οποίος είναι Managing Director για την Ασία και τον Ειρηνικό στην, στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης τον δόκτωρα Άξελ Μπερκόφσκι από το Πανεπιστήμιο της Παβία στην Ιταλία και επίσης Research Fellow στο Ινστιτούτο Πελιστούντι Di Politica του Μιλάνο. Επίσης τον κύριο Μπρούνο Χέλεντορφ, Joint Research Fellow στο ε, Ινστιτούτο Egmont στο Βέλγιο και το Ευρωπαϊκό ε, Κέντρο Πολιτικής. Θα ήθελα να δώσω πρώτα απ' όλα τον λόγο στον κύριο Βίγκαγκ, έτσι ώστε να αναφερθεί σε αυτήν την συμφωνία εταιρική σχέσης με την Ιαπωνία. Έχετε 7-8 λεπτά στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία αυτή. Ε, θα προσπαθήσω να μην ε, ε μιλήσω 8 λεπτά. Απλά θέλω να σας ενημερώσω ότι ε, ε, το Κοινοβούλιο της Ιαπωνίας ε, υπερψήφισε τη συμφωνία αυτή. Θα γίνει η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και στην Ολομέλεια 11 με 13 Δεκεμβρίου ε, ελπίζουμε να γίνει το ίδιο και εδώ στο Κοινοβούλιο ώστε να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιαπωνία, όχι μόνο όσον αφορά την υπογραφή, αλλά και την, όσον αφορά και την κύρωση τη διαδικασία αυτή. Θέλω να σα παρουσιάσω συντομία αυτή την ε, Συμφωνία Στρατηγική Εταιρική Σχέση. Το βασικό σκεπτικό, το βασικό περιεχόμενο, τους βασικούς στόχους και θέλω να συγχαρώ ε, όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά για, αυτή την, ε, για αυτό το έργο. Τον κύριο Πέτριλε που ε, ήταν εισηγητής μας και που ε, τέθηκε επικεφαλής αυτής της διαδικασίας για πολλά χρόνια. Αυτή η νέα συμφωνία δίνει μια πολύ πιο πολιτική διάσταση στην εταιρική μας σχέση. Πολλές φορές ε, πολλοί έχουν την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία συνεργάζονται μόνο σε οικονομικά θέματα, όμως δεν είναι έτσι. Έχουμε μια πλειάδα θεμάτων που μας απασχολούν από κοινού και έχουμε και πολλές κοινέ αξίες που μας δένουν. Μαζί με την οικονομική συμφωνία λοιπόν, η στρατηγική συμφωνία είναι η πρώτη φορά που η Ιαπωνία συνάπτει τέτοιου είδους συμφωνία ε, μια τέτοια στρατηγική συμφωνία που καλύπτει ε, μια τόσο μεγάλη πληθώρα τομέων πολιτικής με εταίρο της. Αυτό βεβαίως θα αναβαθμίσει σημαντικά τις σχέσεις μας με τη χώρα αυτή. Ε, αποτελεί μια ισχυρή βάση για την υπεράσπιση των κοινών αξιών και αρχών μας, αλλά και για την προώθηση της, της υπεράσπιση των κοινών μας συμφερόντων στο διεθνές σκηνικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία είναι ε, εταίροι ε, που ε, συνεργάζονται εδώ και πολλές δεκαετίες στη βάση των αξιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και διμερός αλλά και σε διεθνείς οργανισμούς καθώς και στον τομέα του ελεύθερου εμπορίου. Αυτή η συμφωνία λοιπόν η εταιρική σχέση αποτελεί μια πολύ σημαντική στιγμή σε μια περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας. Γι' αυτό και είναι πιο σημαντική από ποτέ. Με τα νέα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας θα έχουμε την δυνατότητα να ε, επιδιώκουμε ε, κοινή ε, ηγεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας σε μια σειρά από τομείς πολιτικής στο παγκόσμιο στερέωμα. Θεωρούμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε θετικά στη διαμόρφωση, διαμόρφωση της περιφερειακής συνεργασίας, θα μας βοηθήσει στην διεθνή ατζέντα, και η συμφωνία αυτή επίσης καλύπτει και πολλούς νέους τομείς στις διμερείς μας σχέσεις. Στο ΣΠΑ, η, η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, τονώνει και, και ενισχύει τη συνεργασία μας. Βεβαίως η Συμφωνία ε, ελευθέρου εμπορίου που συνοδεύει αυτή τη στρατηγική σχέση είναι και μια, ένας μηχανισμός ε, που ενισχύει ε, τη συνεργασία. Ε, βεβαίως δεν αρκεί να υπογράφονται τέτοιες συμφωνίες, πρέπει στην πράξη να αξιοποιηθούν όλες οι ευκαιρίες που μας δίνει αυτή η συμφωνία. Είναι μια μελλοντοστραφή συμφωνία που ε, δημιουργεί ένα θεσμικό πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να συζητάμε μια σειρά από ζητήματα και ε, ε, μέσω της συμμετοχής ε, και της εμπλοκής του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Όμως, τη διαφορά θα την κάνουμε μόνο αν αξιοποιήσουμε αυτές τις νέες ευκαιρίες που μας δίνει αυτό το νέο πλαίσιο. Υπάρχουν διατάξεις για στενότερη συνεργασία σε βασικά παγκόσμια ζητήματα και θέματα, όπως για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, όπου έχουμε ισχυρά κοινά συμφέροντα και όπου πρέπει να αναλάβουμε δράση. Επίση, η Ιαπωνία είναι πολύ σημαντικό μα εταίρο στην ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια. Μαζί είμαστε οι μεγαλύτεροι συνεισφέροντε στον κόσμο και θέλουμε αυτό να το αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο μέσω τη στενότερη συνεργασία μα. Σε περιφερειακό επίπεδο υπάρχει η σύνδεση μεταξύ τη ευρωπαϊκή ευημερία και τη ασιατική ασφάλεια, που είναι αμφίδρομη. Η ασφάλεια όταν ε, βρίσκεται σε κίνδυνο στην μία άκρη του κόσμου, αυτό επηρεάζει και στον, την άλλη άκρη του κόσμου. Και αυτό βεβαίως ε, τονίζει και τη σημασία ε, της αλληλεξάρτησης που υπάρχει. Αυτό εκφράζεται και στην παγκόσμια στρατηγική μας του 2016. Να σας αναφέρω μόνο την κορατική Χερσόνησο ως ένα παράδειγμα ή την νότια Κινέζικη θάλασσα ως ένα άλλο παράδειγμα όπου ε, αμφότερες οι πλευρές έχουν κοινά συμφέροντα να συμβάλλουν στην ε, επίτευξη και τη διατήρηση της, ε, της ειρήνης, τη διαχείριση των κρίσεων και την εξασφάλιση της παγκόσμιας τάξης μέσω του διεθνούς δικαίου. Μαζί λοιπόν θέλουμε μέσω αυτού του πλαισίου να δημιουργήσουμε μια πολύ στενότερη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας με την Ιαπωνία. Ένας άλλος ε, αντίκτυπος της στενότερης συνεργασίας είναι η συνδεσιμότητα που θα είναι βιώσιμη, ε, φιλική προς το περιβάλλον, ε, θα έχει κοινωνική διάσταση και που θα είναι και οικονομικά αποδοτική. Πάντοτε στη βάση κανόνων και ε, νομικών πράξεων. Και χαιρόμαστε που η Ιαπωνία αποτελεί τον βασικότερο εταίρο μας ε, στον ε, τομέα της συνδεσιμότητας. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος πρόσφατα παρουσίασαν μια στρατηγική για την συνδεσιμότητα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας που έτυχε και τη υποστήριξη του Συμβουλίου, έχουμε πλέον ένα πλαίσιο το οποίο θα μας επιτρέψει να καταστήσουμε τη συνεργασία μας πολύ πιο συγκεκριμένη και απτή στον τομέα αυτό με την Ιαπωνία. Δεν θα μπω σε, στους διάφορους τομείς συνεργασία συνεργασίας και τις επιπτώσεις που θα έχει η συνεργασία αυτή στις κοινωνίες μας και στις οικονομίες μας, αλλά θέλω να επισημάνω τη σημασία που έχουν τα ενεργειακά ζητήματα τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία και στις δύο πλευρές, καθώς και την προώθηση διαπροσωπικών ανταλλαγών συμπεριλαμβανομένων των πολιτών μας. Επίσης, κατοχυρώνεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εφαρμογή ε, της συμφωνίας μέσω των διακοινοβουλευτικών ε, συναντήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας που θα συμβάλλουν σημαντικά στην περαιτέρω διεύρυνση αυτή τη στρατηγική εταιρική σχέση. Αναμφίβολα λοιπόν και οι δύο πλευρέ και η στρατηγική συμφωνία και η οικονομική συμφωνία θα δημιουργήσουν τεράστια ωφέλη για του πολίτε και τι επιχειρήσει μα και στις δύο πλευρές, κινητοποιώντα ε, του διάφορου εμπλεκόμενου και ενδιαφερόμενου φορεί σε αυτή την πολύ περίπλοκη σχέση που έχουμε με την χώρα αυτή. Αυτά είναι τα ωφέλη που θα μας προσφέρει αυτό το νέο πλαίσιο. Ευχαριστώ κύριε Μπερκόφσκι θα μιλήσετε για την πολιτική της Ιαπωνίας στην Ανατολική, ε, Νότιο-Ανατολική Ασία. Έχετε 8 λεπτά. Θα προσπαθήσω ε, να μιλήσω για άλλα θέματα και όχι για το SPA και το EPA ε, και άλλωστε ε, εγώ ακούσατε και ήδη τώρα κάποια στοιχεία. Εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ περισσότερο με την θέση της Ιαπωνίας σε σχέση με τις σχέσεις νοτιοανατολική και την Νότια Ασία. Είναι γεγονός ότι οι Ιάπωνες και λόγω των όσων αναφέρθηκε, ανέφερε και ο κύριος ε, Βίγκεντ προηγουμένως και λόγω της συνδεσιμότητας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια η, ε, η ιαπωνική πολιτική στην Ιωτερική Ασία έγινε πολύ πιο ε, εντατική και έντονη. Η Ιαπωνία συνειδητοποιεί τις ε, συνειδητοποιεί την κατάσταση η οποία δημιουργείται μετά από την εξωτερική πολιτική ε, που χρηματοδοτεί ε, η Κίνα και επομένως έχει αναλάβει δράση και γίνεται όλο και πιο δραστήρια τα τελευταία χρόνια η Ιαπωνία στην ευρύτερη περιοχή. Η Ιαπωνία προτείνει με την Ινδία και την Αυστραλία ε, και τις Ηνωμένες Πολιτείες ποιοτικά προγράμματα ε, δημιουργίας ε, υποδομών και αναλαμβάνει αντίστοιχε πρωτοβουλίε. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, λαμβάνοντα υπόψη και την εσωτερική κατάσταση τη Ιαπωνία το εσωτερικό πολιτικό θεματολόγιο και η αλλαγή στην ε, πολιτική ασφάλεια και άμυνας της Ιαπωνίας ε, μπορεί να εξηγήσει κάποιες από τις αποφάσεις στην εξωτερική πολιτική. Ε, η Ιαπωνία πλέον δίνει στον εαυτό της το δικαίωμα αυτοάμυνας, πράγμα πολύ σημαντικό όσον αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας με άλλες χώρες. Ήδη από το 2014 η Συμφωνία έχει προχωρήσει σε ε, ε, διαφορετική ερμηνεία ε, του συντάγματος και λαμβάνει υπόψη και την των σχετικά με τα θέματα αυτά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, ε, στην εξωτερική πολιτική της Ιαπωνίας, ε, ε, ήδη από το 2013 έχουν ληφθεί κάποιες άλλες διαφορετικές αποφάσεις. Δεν επιτρέπει πλέον η Ιαπωνία στον εαυτό της να εξάγει όπλα και τεχνολογία η οποία σχετίζεται με τα όπλα. και ε, επομένως ε, ε, εντείνεται και η συνεργασία με χώρες της περιοχής αλλά και με την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο κλπ. Και αυτό μπορεί ενδεχομένως να έχει, άμεση, μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στο τι μπορεί η Ιαπωνία να κάνει στην περιοχή. Το 2016 ε, έδωσε δύο πετρελαιοφόρα πλοία στις ε, Φιλιππίνες, καθώς επίσης ε, και πρόσθεσε και το θέμα της ασφάλειας της αεροπλοείας. Επίσης ξεκίνησαν σχέσεις με το Βιετνάμ, όπου δόθηκαν δύο νέα πλοία, ενώ μέχρι τότε δίνοντας το ανόη μονάχα ε, πλοία μεταχειρισμένα από δεύτερο χέρι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, με, την, ε, με τις χώρες που ανέφερα αλλά και με την Ινδονησία μέσω της ίδιας πολιτικής των πλοίων έχουν αναπτυχθεί νέες σχέσεις. Μάλιστα με την Ινδονησία έχει θεσπιστεί ένα θαλάσσιο φόρουμ για την ασφάλεια των θαλασσών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουν κοινούς προβληματισμούς ως όσον αφορά τον ε, επεκτατισμό, τον εδαφικό επεκτατισμό της ε, Κίνας. Ε, αυτή τη στιγμή η Κίνα εξηγεί ένα κείμενο του 1947 για να εξηγήσει την δυνατότητα επέκτασης και διαφοροποίησης των συνόρων και μετακίνηση της Dash Line. Ε, αυτό ε, θεωρείται ότι είναι, θεωρεί η Κίνα ε, ότι είναι δικαίωμά της βάσει αυτού του κειμένου του 1947 και η Ιαπωνία πλέον έχει αναπτύξει νέες αμυντικές στρατηγικές. Επίσης ανοίγεται προς τις χώρες ΑΣΕΑΝ. Οι έξι χώρες της ΑΣΕΑΝ λαμβάνουν πλέον πάνω από το 50% των ελευθέρων συναλλαγών με την Ιαπωνία. Επίσης, πέρσι 110 δις δολάρια δόθηκαν μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας ε, της ε, ΑΣΕΑΝ για ποιοτικές ε, υποδομές έτσι ώστε να εξισορροπηθεί κατά κάποιο τρόπο η πρωτοβουλία της Κίνας για αντίστοιχες επενδύσεις. Βεβαίως όλα αυτά είναι πολύ λιγότερα από όσα έχει βάλει στο τραπέζι η Κίνα. Η επένδυση συνολική της Κίνας στο BBI, BRI ε, φτάνει περίπου στα 4-3. Ε, είναι πολύ λιγότερα μένα, αλλά αποτελούν μια καλή αρχή αυτά που ε, δίνει η Ιαπωνία. Επίσης υπάρχει η λεγόμενη defense diplomacy, η αμυντική διπλωματία της ε, Ιαπωνίας, ε, την οποία χρησιμοποιεί πλέον με την Ασία και ιδίως με την Νοτιοανατολική Ασία. Η Ιαπωνική κυβέρνηση ε, έχει διτή προσέγγιση. Από τη μία πλευρά συνεχίζει την στενή αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πέρα και σε συμπλήρωση αυτό, αυτού, αυτής της πολιτικής έχει νέες θέσεις συνεργασίας με τις χώρες της Ασίας. Επίσης παρουσία στον ειρηνικό ε, είναι όλο και μεγαλύτερη η ε, επιρροή της της περιφέρειας του Ειρηνικού. Ε, έχει λοιπόν η Ιαπωνία δημιουργήσει μια ειδική πολιτική. Κίνα, φεύγουμε, ξεφεύγουμε λίγο, από την Ιαπωνία, αν μου επιτρέπετε, και, να, ε, και από την νοτιοανατολική μάλλον Ασία. Και να πω το εξή: ε, παρά τα προβλήματα που διμερώς υπάρχουν μεταξύ Κίνας και ε, Ιαπωνίας, διότι υπάρχει και μια πάγια ε, και σοβούσα εδαφική αντίθεση μεταξύ των χωρών, γίνεται ε, ε, ε, πριν από μερικούς μήνες έγινε μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών της λεγόμενης Belt and Road Council. Δηλαδή η Κίνα συμφώνησε να συζητάει στο μέλλον τουλάχιστον για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμβάλλει στις καλύτερες σχέσεις στην Belt and Road Initiative. Το Τόκιο ε, μέσω του Πρωθυπουργού Άμπε έχει αναφέρει ότι ε, ενδεχομένως ε, θα ε, επιτρέψει την, την εισαγωγή προγραμμάτων μέσω αυτού του Belt and Road Initiative με κάποιες προϋποθέσεις όμως ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι ισορροπημένα προγράμματα, βιώσιμα προγράμματα και ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να έχει και η Ιαπωνία την δυνατότητα οικονομικής οικειοποίησης των προγραμμάτων μαζί με κάποιες άλλες προϋποθέσεις ε, αυτά είναι πολύ σημαντικό πάντως ε, γιατί ναι, λένε, ε, αναφέρουμε σαφώς ότι είναι σημαντικά θέματα, υπάρχει ένα ξεκίνημα διαλόγου και βεβαίως γνωρίζουμε ότι, και οι προϋποθέσεις, ότι όλες οι προϋποθέσεις που βάζει η Ιαπωνία προφανώς δεν θα καλυφθούν αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι ένα θετικό πρώτο ε, όσον αφορά τώρα την, ε, ε, την συμβολή της Ιαπωνίας σε αυτή την πρωτοβουλία Belt and Road Initiative. Μου δίνετε λίγο χρόνο. Εντάξει, είναι, το δώρο μου για τα γενέθλιά μου, λίγα περισσότερα λεπτά. Η Ιαπωνία και Ινδία. Βεβαίως αυτό ξεπερνάει λίγο την νοτιοανατολική ανατολικη Ασία, μιλάμε για Νότια Ασία. Ωστόσο, όσον αφορά και τις δύο χώρες, την Ιαπωνία και την Ινδία. Ε, η ε, ανατολική πολιτική της Ινδίας, έτσι όπως εγκρίθηκε πριν από δύο χρόνια, ε, έχει επηρεάσει την σχέση με την Ιαπωνία, διότι οπωσδήποτε είναι και η Ιαπωνία μέσα στο κάτω και είναι ακρογωνιαίος λίθος της Act της Ινδίας. Έχει συμφωνηθεί αμυντική συνεργασία με πολύ συγκεκριμένους όρους, ε, κοινέ επιχειρήσεις, κοινέ ασκήσεις μεταξύ της ε, Ινδίας και της ε, Ιαπωνίας, πολλές φορές και με συμμετοχή και της Αυστραλίας. Επίσης, μια συμφωνία η οποία ε, ε, ονομάζεται ACSA και αναφέρεται σε κοινή χρήση λογισμικού ε, στοιχείων και συγκεκριμένη συνεργασία για ασφάλεια και άμυνα επί τόπου. Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Χέλεντορφ τώρα, ο οποίος θα μας μιλήσει για την ΙΟΠ η Ιαπωνία ως παγκόσμιο εταίρο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ για τη χαρά που μου δίνετε να έρθω εδώ και να σας μιλήσω για αυτά τα θέματα. Αυτό το οποίο μένα καταρχήν με ξέπληξε όταν ερευνούσα το θέμα, προσπαθώ τώρα να πέρασω τις διαφάνειες, είναι το πόσο λίγο συζητάμε τις διμερείς σχέσεις με την Ιαπωνία. Υπάρχει η αναθέρμανση Το πλαίσιο είναι λοιπόν τώρα ότι πρέπει να δούμε ένα νέο τρόπο διεθνής πολιτικής και κάτι βασικό ήταν η συνάντηση που έγινε ανάμεσα στους ηγέτες των ΗΠΑ και της Βόρειας Κορέας. Λοιπόν, να σας πω τα εξή σημεία. Πρώτα απ' όλα, ότι βρισκόμαστε σε μια περίεργη στιγμή. Υπάρχει μια ευθυγράμμιση των πλανητών, μπορούμε να πούμε. Αν δεν το είχαμε αυτό, η συνεργασία θα ήταν διαφορετική, όπως ήταν διαφορετική πιο πριν από τότε που άρχισε η συνεργασία από το 2011 που άρχισαν διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, συνέπεια της προσέγγισης αυτής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας είναι τέτοια που δεν πρέπει να ασχοληθούμε μόνο με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις στις σχέσεις μας, αλλά να δούμε και τι άλλες προκλήσεις αντιμετωπίζουμε και οι δύο. Και το επιχείρημά μου είναι ότι δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το εμπόριο που είναι αυτή η συμφωνία εταιρική σχέση, αλλά να κοιτάμε και την εθνική ασφάλεια. Η συνδεσιμότητα, το θέμα του, της κλιματικής αλλαγής, αλλά και άλλα. Πάντως αυτή είναι η τομή σε πάνω στους οποίους πρέπει να έχουμε αποτελέσματα. Και αυτό ακριβώς είναι το επόμενο σημείο μου, ότι πρέπει να έχουμε αποτελέσματα. Δηλαδή δεν πρέπει να αρκούμαστε σε έναν κατάλογο επιθυμιών προτεραιοτήτων, εντάξει δεν μπορούν όλα να είναι προτεραιότητα, πρέπει να περάσουμε και στα αποτελέσματα, τα οποία μπορούμε να αξιολογήσουμε στη συνέχεια ως επιτυχή ή λιγότερο επιτυχή. Τώρα, έρχομαι πάλι το πρώτο επιχείρημα, δηλαδή το κοινό συμφέρον που έχουμε, που ποτέ δεν υπήρχε παλιότερα. Ε, αντιμετωπίζουμε και δύο κοινωνίες οι οποίες γυράσκουν ε, σιγά σιγά. Υπάρχει δηλαδή μια κοινωνική πτυχή και πρέπει να τροποποιήσουμε και τις οικονομίες μας για να πετύχουμε οικονομική ανάπτυξη. Όλα αυτά βέβαια μας ε, ενώνουν μαζί φυσικά. Στην η απορία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολλά κοινά. Το Made in China 2025, για παράδειγμα, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και η ΜΕΝ και η ΔΕ. Και τέλος, ότι αλλάζει το περιβάλλον ασφάλειας. Η Κίνα για την Ιαπωνία. Τα αναφέραμε ήδη. Αλλά επίση και ένα αντιευρωπαϊκό μέτωπο από τη Ρωσία, για παράδειγμα που σίγουρα κάνει τις ζωές μας και τις προπτικές μας πιο δύσκολες, αλλά και μας προσεγγίζει περισσότερο με την Ιαπωνία. Δεύτερον, η προσέγγιση. Πρώτον, έχουμε το Brexit. Θα έλεγα ότι πρόκειται για κάτι που ναι μεν μας αναγκάζει να αντιδράσουμε, αλλά βέβαια από την αρνητική άποψη. Είναι όμως μια προτεραιότητα πρόσβαση στις αγορές, οικονομικές σχέσεις, εμπόριο. Όλα ήταν πιο εύκολα πριν γιατί γινόντουσαν μέσω του Λονδίνου. Τώρα αποχωρεί το Λονδίνο και συνεπώς οι σχέσεις ανάμεσα στις Βρυξέλλες και το Τόκιο δεν είναι πια τόσο εύκολες. Και κάτι άλλο είναι η διεθνής ε, τάξη Τώρα είμαστε σε μια κάπως περισσότερο ασταθή και αβέβαια δεδομένου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά είναι κοινέ προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μαζί. Συνεπώς χρειάζεται να συνεργαστούμε. Όχι μόνο στους τομείς που συνεργαζόμασταν μέχρι τώρα, με ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι τώρα, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα και πρέπει να τα κάνουμε για να στηρίξουμε ένα πολυμερές ε, πλαίσιο κανόνων. Στην πράξη τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Και εδώ δεν πρόκειται μόνο για το ότι πρέπει να δεσμευτούμε για το ένα ή για το άλλο, αλλά είναι ότι μαζί πρέπει να βάλουμε κάτι στο τραπέζι. Και το θετικό της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης είναι ότι πείθει στα λόγια, αλλά τώρα πρέπει να αποδείξουμε ότι πείθηκε στις πράξεις. Πρέπει λοιπόν να φέρουμε αποτελέσματα, τα Benomics στην Ιαπωνία για παράδειγμα, αλλά και εμείς στην Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργήσει υπέρ της Ευρώπης κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρξει επίσης μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Όσον αφορά την διεθνή ασφάλεια θα μπορούσαμε σίγουρα να κάνουμε περισσότερα και πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να προστατεύσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σκεφτεί το, τη δική της ασφάλεια και το βλέπουμε αυτό με το INF με τις προπτικές που δίνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε ότι διπλωματικά και εμείς ε, πρέπει να τονίσουμε τη θέση μας. Υπάρχουν κίνδυνοι για τη μη διάδοση των όπλων, για παράδειγμα. Φυσικά υπάρχουν και πολλά άλλα, ασφάλεια, επιχειρήσεις και σε αυτά πρέπει να συνεργαστούμε. Η ασφάλεια στη θάλασσα Πρέπει να υπάρξει συνδυτοποίηση για την τεχνολογία που διαθέτουμε. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία σήμερα μπορούμε πια να τα δούμε σαν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Επίτα, όσον αφορά την ανάπτυξη και τις υποδομές. Και εδώ θα πρέπει να επιταχύνουμε κάπως με την Ιαπωνία για ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα για συνδεσιμότητα. Είναι ένας αφυσικός εταίρος μας η Ιαπωνία γιατί έχουμε κοινέ αρχές και αξίες. Πρέπει να δούμε πώς θα φτάσουμε στο BRA, το οποίο είναι αναγκαίο, πρέπει να είναι μια επιτυχία και είναι μια βασική στιγμή αυτή. Οι Ιάπωνες θα είναι πραγματιστές, θα προσαρμόσουν τον τρόπο εργασίας τους και στον BRI έχουμε τώρα και εμείς την ευκαιρία. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσω όμως αυτή η ευκαιρία και για την κλιματική αλλαγή πρέπει να συνεργαστούμε επίσης όσον αφορά τη Συμφωνία των Παρισίων μαζί. Θα σταθώ σε αυτά. Το μόνο που έχω να πω ακόμα είναι ότι αυτή η... αυτός ο συντονισμό των πλανητών, αυτή η ευθυγράμμιση των πλανητών δεν θα κρατήσει για πάντα, οπότε πρέπει να υποφεληθούμε τώρα. Και όσο πιο γρήγορα το κάνουμε, τόσο το καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις παρεμβάσεις αυτές. Τώρα να δώσω το λόγο στον ε, κύριο Πέτρελε, τον συγητή μας για τις σχέσεις μας με την Ιαπωνία. you, ε, Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη προσκεκλημένη μας, κύριε Πρέσβη. Είναι μεγάλη τιμή και πρόκληση για εμένα το ότι ανέλαβα τη σύνταξη των εκθέσεων αυτών εδώ και δύο θητείες σχεδόν. Ο κόσμος ε, έχει αλλάξει πολύ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεών μας. Όμως βλέπω ότι με τις κοινέ μας προσπάθειες έχουμε καταλήξει στο τέλος μιας πολύ απαιτητικής διαδικασίας μέσω της οποίας καταφέραμε να ενισχύσουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ δύο παγκόσμιων εταίρων. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι δεν έχουμε μόνο κοινά συμφέροντα, αλλά και κοινέ φιλοδοξίες να οικοδομήσουμε μια βιώσιμη εταιρική σχέση, η οποία είναι δυνατή μόνο στο βαθμό που βεβαίως ε, συμμεριζόμαστε κοινέ αξίες και αρχές. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει. Στην αρχή υπήρχε μια καλή διάθεση, αν θέλετε, μια συμπάθεια. Πλέον όμως βρισκόμαστε σε απόλυτο συντονισμό όσον αφορά την προστιθέμενη αξία που έχει αυτή η διαδικασία, η κοινή που ακολουθούμε. Και τα λέω αυτά γιατί ε, και μένω σε αυτά, ε, διότι θα μου ζητήσετε από ό,τι ξέρω και τον, να, να κάνω κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Τώρα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο από τους ισολογιστές, τον κύριο Καν, ο οποίος αν κατάλαβα καλά θα παρουσιάσει αυτό που είχε ετοιμάσει ο Ντέιβιντ Μάρτιν, γιατί ο Ντέιβιντ Μάρτιν είναι σκιώδης για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπεργκόφσκι, καταρχάς χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρέσβη, παίρνω το λόγο εκ μέρους του κύριου Ντέιβιτ Μάρτιν, που είναι σκιώδης εισηγητή για τις ε, στρατηγικέ εταιρικέ σχέσει μα εκ μέρου της ομάδας μας. Δυστυχώ δεν μπορεί να είναι εδώ. Υποστηρίζει την SPA γιατί θα ενισχύσει τι πολιτικέ μα σχέσει με την Ιαπωνία και θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο για τον τακτικό διάλογο, τη συνεργασία σε διάφορα σημαντικά ζητήματα όπω είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από αυτή την άποψη ο Ντέιβιτ θέλει να ρωτήσει τον εκπρόσωπο της ε, ε, υπηρεσία εξωτερική δράση για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την θανατική ποινή. Βρισκόμαστε σε συνεργασία και διάλογο για αυτό το θέμα. Θα μας δώσει η Στρατηγική Συμφωνία τη δυνατότητα να ασκήσουμε πίεση στην Ιαπωνία για να προβεί στην κατάργηση της θανατικής ποινής. Στο πλαίσιο της Οικονομικής ε, Συμφωνίας, εμείς ε, ασκούμε πίεση στην Ιαπωνία να κυρώσει δύο συμβάσεις του ILO για τις διακρίσεις και την καταναγκαστική εργασία. Ε, θεωρούμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί και μια ε, ε, μάλλον όχι, θεωρούμε σημαντικό το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί και μια δημιουργική, ομάδα εργασίας για αυτά τα θέματα. Δεύτερον θέμα, ε, το θέτει αυτό το θέμα η, η, η Ευρωπαϊκή ε, Υπηρεσία εξωτερική δράση στην Ιαπωνία. Άλλο θέμα, πειράματα σε ζώα γίνονται στην Ιαπωνία απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχούν για αυτή την πρακτική. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του Μαρτίου, το 89% των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει περισσότερα πράγματα για την ενίσχυση και την προώθηση τη ευημερία των ζώων στον κόσμο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίση έχει εγκρίνει ψήφισμα για την απαγόρευση των πειραμάτων σε ζώα για καλλιτικά προϊόντα. Έχετε θέσει αυτό το ζήτημα στην Ιαπωνία. Γιατί εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτήν την στρατηγική συμφωνία για να προωθήσουμε την ενωσιακή πολιτική για την ευημερία των ζώων στην Ιαπωνία. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος, λέει ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω τι να κάνουμε τώρα. Θέλει κάποιος από εσά να μιλήσει ε, ε, σε σχέση με αυτά που είπαν ε, οι βουλευτές που μίλησαν προηγουμένως. Ωραία. Θα απαντήσω στα θέματα που τέθηκαν στο βαθμό που μπορώ βεβαίω και στο βαθμό που μου το επιτρέπουν οι γνώσει μου. Όσον αφορά τη θανατική ποινή, που είναι μια προφανής διαφορά που έχουμε με την Ιαπωνία, και που δεν είναι και η μοναδική, ξέρετε. Δεν είναι επίση η Ιαπωνία ο μοναδικός ε, στενός εταίρο μας με τον οποίο έχουμε αυτή τη διαφορά. Υπάρχει αυτή η διαφορά ε, και με άλλες δημοκρατίες και άλλα κράτη ε, που ακόμη δεν έχουν αναλάβει βήματα για την κατάργηση της, ανθρώπιν, της θανατικής ποινής, την οποία εμείς βεβαίως υποστηρίζουμε πλήρως την κατάργηση. Εμείς αντιτιθέμεθα στην χρήση θανατική ποινή σε όλες τις περιστάσεις, σε όλες τις περιπτώσεις, θεωρώντα ότι είναι μια απάνθρωπη μέθοδος και ε, λόγω του γεγονότος ότι δεν μπορεί ποτέ κανείς να αποκλείσει ε, την ε, δικαστική πλάν Γι' αυτό και είναι σημαντική και απαραίτητη η της θανατική ποινή για την ε, προστασία τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Έχουμε αναλάβει πολλέ κινήσει προς αυτή την κατεύθυνση ε, ιδίως τις φορές που ε, εφαρμόζεται το μέτρο της θανατικής ποινή στην Ιαπωνία και το χρησιμοποιούμε και το επαναφέρουμε αυτό το θέμα στον πολιτικό μας διάλογο με το Τόκιο. Συστηματικά λοιπόν καλούμε τις Ιαπωνικές αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπιση ενός μορατόριου τουλάχιστον για την θανατική ποινή, κάτι που κάνουμε και στις συζητήσεις μας με άλλους εταίρους μας που εφαρμόζουν τη θανατική ποινή και ε, προωθούμε μια ειλικρινή, ανοιχτή δημόσια συζήτηση, που βεβαίω δεν μπορεί να γίνει υπό την αιγίδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητούμε όμω από τι Ιαπωνικέ Αρχέ να δημιουργήσουν εκείνον τον ε, χώρο, ώστε να γίνει μια ανοιχτή, ειλικρινή συζήτηση στην κοινωνία τη Ιαπωνία, προκειμένου να κατευθυνθεί και αυτή η κοινωνία ε, μακριά από την θανατική ποινή. Αντίστοιχε κινήσει βεβαίω αναλαμβάνουμε και με τι ΗΠΑ. Δεύτερο θέμα πρέπει να σας ομολογήσω ότι το θέμα αυτό δεν ε, καλύπτεται άμεσα από καμία από τις διατάξεις, εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον. Σίγουρα όχι στην στρατηγική συμφωνία εταιρικής σχέσης που ξέρω ε, και που κατέχω το περιεχόμενό της. Φαντάζομαι όμως ότι ούτε στην ε, οικονομική συμφωνία υπάρχει κάτι τέτοιο. Εδώ πρόκειται για ένα θέμα το οποίο βεβαίως μπορούμε να επαναφέρουμε στις συζητήσεις μας με τις Ιαπωνικές Αρχές ε, στη βάση της πολιτικής που ακολουθείται στον τομέα αυτό στη χώρα τους. Τρίτο θέμα ε, που θέσατε είναι η συμβάση του Διεθνούς ε, Οργανισμού Εργασίας. Εδώ υπάρχουν σαφείς δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Οικονομικής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και θεωρώ ότι το στοιχείο αυτό, το θέμα αυτό θα διαδραματίσει, διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις συζητήσεις μας με τους Ιάπωνες εταίρους μας, το οποίο βεβαίως θα πρέπει να ε, συνοδευτεί και από ε, εφαρμοστικά μέτρα στο εσωτερικό της χώρας. Είναι και αυτό ένα στοιχείο της νέας γενιάς εμπορικών συμφωνιών που υπογράφουμε πλέον με διάφορες πλευρές ε, και διάφορες χώρες του κόσμου. Αναφέρομαι κυρίως στη στρατηγική συμφωνία εταιρική σχέση, αλλά βεβαίως αυτά που λέω αφορούν και την οικονομική συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλέσω ε, τον πρέσβη της ε, ε, Ιαπωνίας να πάρει το λόγο. εξοχώτης παρακαλώ έχετε το λόγο. Um, oh, uh, uh, Mr. Chair, thank you very much for... Um, Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την δυνατότητα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις ε, με την ευκαιρία της ακρόασης. Κυρίως θα ήθελα ε, να ευχαριστήσω και τον Προεδρεύοντα ε, και τα μέλη της, Επιτροπής ΑΦΕΤ αλλά και τους ομιλητές. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία σημεία. Κάτι που ανέφερε και ο κύριος Βίγκαντ προηγουμένως. Η, αυτή η συμφωνία εταιρικής σχέσης ε, πραγματικά ενδυναμώνει την εταιρική μας σχέση και την αποφασιστικότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις, όχι μόνο διμερείς, αλλά ε, και τις ε, προκλήσεις που έχουμε απέναντί μας, όπως κλιματική αλλαγή, μεγαλύτερη ασφάλεια, διαχείριση της ασφάλειας, ε, ε, το θέμα της, του εκδημοκρατισμού της Βόρειας Κορέας κλπ. Όλα αυτά τα πιεστικά ε, και σημαντικά ζητήματα και πιστεύω ότι μέσω αυτής της συμφωνίας θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα καλύτερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας. Δεύτερον, όπως είπε και ο κύριος Βίγκαντ, μέσω της ε, συμφωνίας θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ε, ένα καλύτερο και πιο στέρεο νομικό υπόβαθρο για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Ιαπωνίας. Δεύτερον, ο τρίτος ομιλητής, ο κύριος Χέλντεντορφ, αναφέρθηκε σε κάποιους εξωγενείς παράγοντες που οδηγούν σε αυτή την προσέγγιση στο ραπροσμό. Να πω ότι συμφωνώ με τις αιτιάσεις του, αλλά αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες πιστεύω ότι όθησαν ε, ε, προς το leadership της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μονάχα το leadership της ε, Ιαπωνίας. Νομίζω ότι αυτή η αίσθηση επίγοντος, η αίσθηση της κρίσης μας υποχρέωσε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της Συμφωνίας Εταιρικής Στρατηγικής Συνεργασίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το τρίτο, αυτή η πρωτοβουλία BRI. I'm counterbalancing BRI. I'd rather not use... Ε, αυτό το Belt and Road Initiative είναι τόσο... Even before the BRI was... Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Then of course, uh, also, of course, I think um, we, we believe... I... Βεβαίως, βεβαίως πιστεύουμε ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Νέα Ισλανδία, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ινδία. Πραγματικά αναγνωρίζουμε όλοι την σημασία ε, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των αξιών που συνδέονται με τον άνθρωπο. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία άρρηκτα συνδέονται με, την, με τη σχέση μας. Και μέσω της συμφωνίας θα δοθεί μεγαλύτερη ενδυνάμωση ε, και όθηση στις ε, σχέσεις μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη. Ο κύριος Δαρκόφσκι τώρα. Ο κύριος Μπερκόφσκι. Ναι, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για τις ε, παρατηρήσεις σας. Βεβαίως, η συμφωνία, η αρχική με την Ιαπωνία είναι παλιότερη από το 2006. Όταν τα κοιτάμε όλα αυτά και θα είμαι ειλικρινής, γιατί δεν είμαι πολικός ούτε διπλωμάτης, είμαι ακαδημαϊκός, ο τρόπος που αντιμετωπίζεται η συνεργασία στην Αυστραλία, στις Ηνωμένε Πολιτείες, στον Ειρηνικό για το σύνολο, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι το αντίθετο από αυτά που κάνει η Κίνα στην περιοχή με την εδαφική της πολιτική και τους εδαφικούς ισχυρισμούς της. Και πολλά από τα σχέδια μέσα στην BRA έχει να κάνει με το τι κάνουν και οι τέσσερις χώρες. Είτε πρόκειται για μία αντιπρόταση παραγωγική, είναι μια αντίδραση στα όσα κάνει από το 2013 η Κίνα η οποία συνδέει την Ασία με την Ευρώπη μέσω της πρωτοβουλίας «Μία ζώνη, ένας δρόμος». Κάποιες από τις πολιτικές, οι πολλές από τις πολιτικές της Κίνας, στην νοτιοανατολική Κίνα, δεν ακολουθούν τους διεθνείς κανόνες. Για παράδειγμα, η Κίνα δεν έχει πρόβλημα να γνωρίσει το διεθνές δίκαιο, την απόφαση της διαιτησίας το 2016. Το δικαστήριο είχε πει ότι το νησί στα πλαίσια της περίφημης dash line, της διαχωριστικής γραμμής, δεν αποτελεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Έτσι είπε το δικαστήριο. Το γνώρισε η Κίνα. Οι δημοκρατικές χώρες όμως στην περιοχή έτσι έχουν μια ευκαιρία να ενωθούν και να προτείνουν κάποιο αντίβαρο. Κλείνει το μικρόφωνο του ομιλητής. Οι προσπάθειες της Ιαπωνίας να κάνει κάτι πρέπει να αποδώσουν. Πρόεδρος, ευχαριστώ και μια σύντομη αντίδραση, παρακαλώ και από εσά. Ναι, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ. Εξοχότατε. Ακριβώς αυτό Ανούσα και εγώ ότι αυτή η προσέγγιση τώρα προσμό δεν είναι μόνο από την Ιαπωνία η οποία θα έρθει στις Βρυξέλλες, πρέπει να είναι και από τις δύο πλευρές. Αλλά ακριβώ το ότι είναι και από τις δύο πλευρές και με ένα τέτοιο βηματισμό, με ένα τέτοιο ρυθμό που φτάσαμε σε μια ισχυρή συμφωνία όχι μόνο εμπορική αλλά και πολιτική και ίσως και διαχειρισμού του μόνο αργότερα είναι κάτι μοναδικό που δεν είχαμε δει για πολλά χρόνια υπήρχε μια απόσταση, αλλά πάντα είχαμε καλές σχέσεις. Χρειάστηκε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον έτσι ώστε και οι Βρυξέλλες και η Ιαπωνία να αντιληφθούν πόσο φυσική σύμμαχοι και εταίροι είναι. Δεν έχουν μόνο κοινά συμφέροντα, αλλά και κοινέ αρχές και αξίες. Και έτσι είτε πρόκειται για τη διάδοση των όπλων, είτε πρόκειται για την ε, κυβερνοασφάλεια, είτε πρόκειται για το κράτος δικαίου. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία διπλωματικά συζητιούνται, αλλά τώρα υπάρχει και πολιτικά ανστερνισμός. Και αυτό ακριβώς εννοούσα. Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου είναι ένα πρόβλημα για όλους βέβαια και κυρίως για την Ιαπωνία, ακριβώς για το καθεστώς των νησιών εκεί. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε μία τάξη που να βασίζεται ε, σε διεθνείς συμφωνίες. Και βάσει αυτού θα αξιολογηθεί και η συμφωνία αυτή Ευρώπης-Ιαπωνίας. Πρόεδρος, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταίος, που θα πάρει το λόγο στην ακρόασή μας εδώ είναι ο Άλης Πέτερλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως εισηγητής για την συμφωνία αυτή στρατηγικής σχέσης πρέπει να ευχαριστήσω για τα σχόλια που άκουσα από τους προσκεκλημένους και τους συναδέρφους. Και οι δύο συμφωνίες θα πάρουν χρόνο για να φτάσουν σε ένα νέο στρατηγικό επίπεδο προς όφελος των πολιτών εκατέρωθεν. Πρόκειται για δύο οικονομίες που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο και δύο δημοκρατίες που μοιράζονται την ίδια αντίληψη για την εμπορική συνεργασία. Μέσα στην συνολική ατμόσφαιρα στην οποία ζούμε είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοιου είδους συνεργασία η SPA ενισχύει τη συνεργασία μας θέτοντας τις νομικές βάσεις για ομιακή και άλλη συνεργασία για θέματα τα οποία είναι αμοιβαίως συμφέροντος στα πλαίσια περιφερειακών και διεθνών προκλήσεων. Είναι μια διμερής συμφωνία και συνεργασία η οποία ανοίγει δυνατότητες και για συνεργασία σε άλλους ε, τομείς. Πάνω από 40 τομείς έχουν εντοπιστεί από την κυβερνοσφάλεια μέχρι την υγεία. Για κάποιον λοιπόν, ο οποίος είναι αφοσιωμένος στο έργο μας, θα ξέρετε ότι είναι η πρώτη φορά που το θέμα υγείας συμπεριλαμβάνεται σε μια τέτοια συμφωνία, ώστε να υποφεληθούμε από την τεχνολογία στην υγεία και ενισχύοντας τη συνεργασία μας σε αυτό το τομέα, ενισχύουμε και τη θέση μας στην παγκόσμια αγορά, και βοηθούμε τη, να λυθούν τα προβλήματα υγείας παγκοσμίω από την κοινή μας πραγματογνωμοσύνη. Πιστεύω ότι πολύ θα αποφεληθούμε από μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ μας. Τώρα ο καθηγητής Μπερκόφσκι και ο πρέσβης, η εξοχότης του, αναφερθήκατε στην Ινδία. Θα ήθελα το πνεύμα το οποίο υπερίσχυσε στις διαπραγματεύσεις μας με την Ιαπωνία και η φιλοδοξία μας εκεί να υπερισχύσουν και στις διαπραγματεύσεις μας με την Ινδία που είναι επίσης ένα σημαντικός μας εταίρος. Χαίρομαι που μπορούμε να συμφωνήσουμε και για τον ρόλο των δύο κοινοβουλίων. όταν θα έχει κυρωθεί συμφωνία και τεθεί σε εφαρμογή. Τα δύο κοινοβούλια θα έχουν υπεύθυνο ρόλο και στο μέλλον. Την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο θα ψηφίσουμε και για τις δύο συμφωνίες. Δεν πρόκειται μόνο για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, πρόκειται για συμφωνία μεταξύ ισότιμων εταίρων, οι οποίοι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν από κοινού προκλήσεις και να φροντίσουν να υποφεληθούν αμοιβαία περιμένουμε να στηριχθούν ευρέω και οι δύο συμφωνίες. Και έτσι να αρχίσουμε γρήγορα συνεργασία με τους Ιάπωνες εταίρου. Μπαίνουμε σε ένα νέο στάδιο. Είναι μια νέα πρόκληση. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για φιλόδοξη εφαρμογή των δύο αυτών συμφωνιών. Τέλος, Ευχαριστώ πολύ την διαπραγματευτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Το ίδιο θέλω να πω και για τους σκιώδες συζητητής και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την εξοχότητά του και τον προκάτοχό σας που έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά προκειμένου να στηρίξει την διαδικασία αυτή. Εκφράζω και την ευγνωμοσύνη μου σε πολλούς συναδέρφους που δεν είναι εδώ σήμερα, αλλά η απουσία τους είναι καλό σημάδι. Έτσι θέλω να το ερμηνεύσω. Γιατί η αίθουσα είναι γεμάτη όταν έχουμε να κάνουμε με προβλήματα. Εδώ δεν υπάρχουν προβλήματα. Έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ και για τις παρατηρήσεις και για τη συνεργασία. το έργο μας θα στεφθεί με επιτυχία, ελπίζω πολύ σύμφωνα. Αρικατό, λέει ο Πρόεδρος. Ωραία. Αρικάτο και από μένα λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα λάβει χώρα τη Δευτέρα στο Στρασβούργο στις 7.30 ε, το απόγευμα μαζί με την ΔΕΒΕ. Θα έχουμε και τον κύριο Σεντσόφ ε, του βραβείου Ζαχάροφ. Ευχαριστώ.